να ψηφίσουμε δηλαδή και να υιοθετήσουμε την θέση μας για τον προϋπολογισμό Τώρα, η επόμενη συζήτηση που ακολουθεί δηλαδή είναι μια συζήτηση ανάμεσα στους σκιώδεις συζητητές, αλλά χρησιμοποιούμε την μετάφραση των τους διερμηνείς δηλαδή για να κάνουμε αυτή τη συνεδρίαση και θα πρέπει δηλαδή να φύγετε αμέσως όλοι μετά. Ε, για θα ξανασυνεχιστεί η συνεδρία των συντονιστών η οποία δεν τελείωσε. Να σας κάνω κάποιες ανακοινώσεις ενημερωτικές. Είχαμε μια πρώτη συνάντηση τριμερή τριμερούς διαλόγου για την κρίσιμη αυτή πρόταση για τις καθυστερημένες πληρωμές ε, και νομίζω ότι κάνουμε κάποια πρόοδο. Αυτό λοιπόν προς ενημέρωσή σας και για να ξέρετε ότι σύμφωνα με τις εργασίες αυτής της Επιτροπής, συνεχίζοντάς τις, προσπαθούμε να κινηθούμε προς μια λογική συμφωνία που θα ωφελήσει τις ΜΜΕ και δεύτερον να σας πω ότι θα γίνει μια σημαντική συνεδρίαση εκτός από τις επιτροπές, αλλά μας δίθηκε να την υποστηρίξουμε στις 14 Οκτωβρίου. Γενικός Γραμματέας του Κοινοβουλίου επέτρεψε τη χρήση των χώρων του Κοινοβουλίου από την Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Πανεπιστημίων που προσπαθεί να συνδυάσει τη διαδικασία της Μπολόνια για τις ε, επαγγελματικέ ε, τα επαγγελματικά πτυχία και την αναγνώριση, αμοιβή αναγνώριση αυτών. Αυτό συνδέεται με τη δουλειά της Επιτροπής μας ε, για την εξέταση του ισχύοντος κανονισμού, του καθεστώτος μάλλον για την αναγνώριση των ε, πτυχίων. Ε, να σας ενημερώσω ότι πήγα επίσης σε μια αποστολή ως πρόεδρος της Επιτροπής μας στην Ουάσιγκτον τον Ιούλιο, όπου είχα εξαιρετικά χρήσιμες και θετικές επαφές σε ψηλού επίπεδο με αρκετούς επιτρόπους, μάλλον προέδρους επιτροπών του Κογκρέσου, που έχουν, απασχολούνται με την προστασία του καταναλωτή, την τυποποίηση και θέματα αγοράς. Και επίσης είχα επαφές με την ε, Αμερικανική κυβέρνηση και μπόρεσα να ανανεώσω την γνωριμία μου με τον πρόεδρο της Επιτροπής, ε, της Αμερικανικής Επιτροπής για την Ασφάλεια των Προϊόντων που ήρθε στην Επιτροπή μας τον Ιούνιο και μάλιστα είχα και ένα γεύμα με όλα τα μέλη της Επιτροπής της, με βοήθησαν πολύ, μου ε, κάνονταν άλλες συναντήσεις ε, και είχαμε και συναντήσεις στο Υπουργείο Εμπορίου Μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον ε, των ζητημάτων και το θέμα της τυποποίησης στο πλαίσιο της διεθνούς αγοράς και του διεθνούς εμπορίου είναι κάτι το οποίο θα προκύπτει διερκώ στην ημερήσια διάταξη και νομίζω πως πολλοί έχετε στις επαφές σας με τη ΣΥΠΑ και άλλες χώρες ε, τέτοιου είδους συζητήσεις θα μπορούσατε ίσως να παρακολουθήσετε το θέμα. Μεγάλη επιτυχία η επίσκεψη λοιπόν. Ελπίζω να είχατε εξίσου παραγωγικές και αναπαυτικέ. Ε, ε, διακοπές. Να σας πω ότι επίτροπος με τον, οι επίτροποι μάλλον με τους οποίους συνεργαζόμαστε διακαώς επιθυμούν να μας συναντήσουν. Χθε είχα μια συνάντηση με τον νέο Γενικό Διευθυντή της Γουδού Αγορά τον κύριο Τζόνας Μπλουμ που είναι επίσης ε, ε, πρόθυμος να συνεργαστεί μαζί μας και ψάχνουμε να βρούμε μια ευκαιρία να έρθει να μας ε, δει εδώ στην Επιτροπή μας μέσα στο φθινόπωρο. Η συνεργασία μας λοιπόν καλά κρατεί με την γάμα δέλτα αγορά. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε στην ψηφοφορία την έκθεση της κυρίας Ρούλε και ονόματος της Επιτροπής για τον προπολογισμό. Έχουμε συζητήσει και πρέπει τώρα να το ψηφίσουμε. Θα δώσω την κυρία Ρούλε την ευκαιρία να μας πει, ε, να μας πει πού βρισκόμαστε με τις ψηφοφορίες. Και πού βρισκόμαστε και με τον προπολογισμό. Η κυρία Ρούλε, θα είμαι πολύ σύντομη. Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα για την πολύ καλή συνεργασία με τους κοιόδης εισηγητές που ήταν πρόθυμοι, παρότι είχαμε διακοπές, να δούνε για άλλη μια φορά τις ε, τροπολογίες και να δεχθούν τις πιεστικές προθεσμίες. Και θέλω επίσης να ευχαριστήσω και την Γραμματεία για την ε, υποστήριξη κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών. Να υπάρξει η δουλειά, να καλυφθεί έργο ε, για τον προπολογισμό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ευχαριστώ για την υποστήριξη και βοήθεια. Σε πρώτη γραμμή θέσαμε το στόχο μας τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, να τα μπορέσουμε να τα διασφαλίσουμε. Ξέρετε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε δύσκολες διαπραγματεύσεις και με την κρίση στα κράτη-μέλη, δημοσιονομική οικονομική κρίση και η υποστήριξη όλων των σχεδόν εισηγητών ώστε να μεριμνήσουμε ότι τα κονδύλια που είχε εγγράψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αποκατασταθούν και να διασφαλιστούν και ότι οι περικοπές του Συμβουλίου θα αντιμετωπιστούν. Σε ένα σημείο κάναμε μια μικρή εξαίρεση στο Solvit. Έχουμε μια ξεχωριστή γραμμή ως κονδύλιο που υποστηρίζεται για το Solvit και βρισκόμαστε κάπως κάτω από το όριο και ελπίζουμε ότι θα βρεθεί η υποστήριξη της Επιτροπής Προϋπολογισμών ώστε το κονδύλιο για το Solvit να εγκριθεί Στη συνέχεια στην ψηφοφορία νομίζω μπορούμε το σύνολο αυτό των προτάσεων να το ψηφίσουμε μέχρι το ψήφισμα. Στο ψήφισμα υπάρχει ένα σημείο το οποίο είναι αντιφατικό, είναι αμφίσιμο. Υπάρχει μια τροπολογία του κυρίου Ντε Γιόγκ που δυστυχώς δεν μπορώ να την υποστηρίξω διότι θεωρώ ότι είναι πολύ γενικόλογη και δεν ανήκει στον τομέα των δημοσιονομικών για τον προϋπολογισμό. Προσπάθησα σε όλα τα σημεία και στο ψήφισμα ακόμα την αρμοδιότητα της ΙΝΚΟ, της δικής μας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, να την σεβαστούμε και να μην ξεπεράσουμε τα εσκαμμένα της αρμοδιότητες μας, για να έχουμε καλές πιθανότητες να πετύχουμε τους στόχους μας. Ευχαριστώ. Uh, well, thank you very much indeed for your very... εγώ σας ευχαριστώ για όλο το έργο σας που ήταν πολύ εμπεριστατωμένο και ας δούμε τώρα τον κατάλογο ψηφοφορίας που είναι χωρισμένο σε δύο μέρη. Έχουμε όλες τις γραμμές του προπολογισμού και η συγκίτρια συστήνει να υποστηρίξουμε όλες τις προτάσεις για τις γραμμές του προπολογισμού και έχουμε το ψήφισμα όπου θα ψηφίσουμε για τις παραγράφους. Εγώ θα ήθελα να ξέρω από τις πολιτικές ομάδες Μπορούμε να βάλουμε όλες τις γραμμές του προπολογισμού unblock, να τις ψηφίσουμε ή θέλετε να ψηφίσουμε χωριστά μία-μία. Όχι, unblock. Πολύ ωραία. Ψηφίζουμε λοιπόν τότε για όλες τις γραμμές του προϋπολογισμού που έχετε στο σχέδιο 6.750 μέχρι 6.755. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, εγκρίνονται ομόφωνα. Και τώρα πάμε στο κομμάτι του ψηφίσματος. Εδώ θα ψηφίσουμε χωριστά. Παράγραφος 2. Τροπολογία Σόντεργαρντ και Ντεγιόγκ. Υπέρ κατά απορρίπτεται παράγραφος 5 ρούλε υπέρ κατά εγκρίνεται παράγραφος 6 υπέρ κατά εγκρίνεται παράγραφος 7 υπέρ κατά εγκρίνεται Ψηφίζουμε λοιπόν για το σύνολο της νομοδότησης ε, για τον προπολογισμό υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. Να διάποχες και μια ψήφο κατά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Ρούλε. Ξέρουμε ότι είστε εσείς ο σταθερό μας εκπρόσωπος της διαπραγματεύσης του για τον προπολογισμό. Τέλος λοιπόν αυτής της συνεδρίασης τώρα.